Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης ε, που προβλέπει τις παρεμβάσεις ενός λεπτού με βάση το άρθρο 163 του κανονισμού. Το λόγο πρώτο ο κύριος Στέφανετς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι πολύ σοβαρό θέμα και οι συμπολίτες μας περιμένουν αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης ε, της τρομοκρατίας. Επίσης, περιμένουμε επιτέλους την πρόταση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, πρέπει να έχει καλύτερη επικοινωνία με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες, γιατί κάποια, κάποιες παράγραφοι της ε, νέας οδηγίας θα παραβιάσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας, νομίζω, των συμπολιτών μας. Θα πρέπει να προβλέψουμε διασύνδεση των εθνικών μητρών, αλλά δεν θα πρέπει να τιμωρούμε νομοταγείς πολίτες. Θα πρέπει να κάνουμε κάποια διαφοροποίηση και δεν θα πρέπει με τα νέα μέτρα να αυξηθεί ο αριθμός ε, των ε, παράνομων κατόχων πυροβόλων όπλων. Μάλιστα, χαίρομαι που εκπρόσωποι Σλοβενικής Οργάνωσης ε, κατόχων όπλων μπόρεσαν να έχουν ακρόαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσουν τις απόψεις. Ο κύριος Τάλι. Θα ήθελα να συγχαρώ τους πολίτες της Σερβίας που στις πρόσφατες εκλογές ε, διατράνωσαν ε, την επιθυμία τους για ένα φιλοευρωπαϊκό και ευρωπαϊκή πορεία της ε, Σερβίας, της πατρίδας τους. Θα πρέπει έτσι η Σερβία να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενταχθεί η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσει τους πολίτες. Επίσης και οι Ούγγροι της Βοηβοδίνας ε, είχαν πολύ καλά αποτελέσματα και έτσι θα βοηθεί η Ουγγρική μειονότητα να κρατήσει την ισχυρή της εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα. Τους τελευταίους μήνες η Σερβική κυβέρνηση άνοιξε τα πρώτα κεφάλαια των ανταξιακών διαπραγματεύσεων. Επίση, διαπιστώνουμε την δέσμευσή του ε, να αντιμετωπίσουν την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και να ενισχύσουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Τώρα ε, απομένει στα θεσμικά όργανα να κάνουν το δικό του έργο. Γι' αυτό θα πρέπει η Κομισιόν και η, Ευρωπαϊκή Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξουν εκκρεμή κεφάλαια και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 23 τη διαπραγματεύση. Ευχαριστώ. Κύριο Μπουσόη. Ευχαριστώ. Πέρασαν πάνω από πέντε μήνες που οι υπηρεσίες προστασίας παιδιών της Νορβηγίας πήγαν πέντε παιδιά μια οικογένειας παρά τις εκκλήσεις που έχουν γίνει από την κοινωνία των πολιτών και οργανώσεις προστασίας του παιδιού, τίποτα δεν έχει γίνει στη πρακτική της Νορβηγίας. Είναι απαράδεκτο επίσης, στον 21ο αιώνα, ένα βρέφος τριών μηνών αφαιρείται από την οικογένειά του, να το στερείται η οικογένειά του με βάση μια διοικητική απόφαση, ούτε καν διαδικαστική, που μάλιστα στη συνέχεια κυρώθηκε και το παιδί επέστρεψε στου γονείς του. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο και πολύ τραυματικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πιο ρητά και κατηγορηματικά να επισημάνει αυτά τα προβλήματα στη σχέση με την Νορβηγία. Ο κύριο Καπούτο. Grazie, Presidente. È recentemente una... Δημοσιώθηκε πρόσφατα ένας κατάλογος κάποιων τροφίμων τα οποία είναι μολυσμένα και δεν μπορούν να εισάγονται στην χώρα μου. Σαν παράδειγμα κάποια πορτοκάλια από την Αίγυπτο, μαϊντανός από την Ινδία, άλλα προϊόντα από, από την Δομινικανή Δημοκρατία όπως και η μέντα από το Μαρόκο θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τοξίνες που μπορεί να προκαλέσουν και καρκίνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τους ελέγχους εισαγωγής των τροφίμων έτσι ώστε όλα τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να κυκλοφορούν με κάθε δυνατή ασφάλεια. Πολλές φορές τα προϊόντα αυτά παράγονται ε, μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικού και οικονομικού dumping. Ε, και θα πρέπει να υπάρξει φυτοϊγειονομικός έλεγχος εκεί όπου απαιτείται. Θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει τις εισαγωγές πρώτων υλών έτσι ώστε όλοι ε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουν τι επικίνδυνα προϊόντα εισάγονται. Ο κύριος Μαριάς. Ε, όπως ανέφερα και σε προηγούμενη σημερινή συζήτηση, η ηγεσία του ενίσα εδώ και χρόνια μεθοδεύει την απαξίωση της δραστηριότητας του οργανισμού στο ηράκλειο της κρήτης. προώθησε λοιπόν τη διάσπαση του οργανισμού σε δύο κέντρα ένα διοικητικό κέντρο στο ηράκλειο το οποίο πλέον υπολειτουργεί με δέκα υπαλλήλου ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του οργανισμού εργάζεται στο επιχειρησιακό κέντρο που λειτουργεί στην αθήνα. στόχο η πλήρη απαξίωση τη λειτουργία του οργανισμού στο ηράκλειο τη κρήτη και η εν συνεχεία μεταφορά τη έδρα του ενίσα εκτό ελλάδα να γνωρίζει η ηγεσία του ενίσα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να φύγει η έδρα του οργανισμού από το ηράκλειο. θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μαζί με τους τοπικούς φορείς της κρήτης όπως το κάνουμε με συνέπεια ήδη από το 2012 όταν ήμουν βουλευτής ηρακλείου. έδρα του ενίσα είναι και θα παραμείνει η κρήτη ό,τι και αν θέλει η ηγεσία του ενίσα που ήρθε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με αλαζονικό ύφος για να ηρωνευτεί τους ευρωβουλευτές για τον λόγο αυτό και δεν πρόκειται αύριο να εγκρίνω την απαλλαγή του ενίσα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 1312 γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν υπερήφανα τον τίτλο προστατευμένης ονομασίας προέλευσης. Είναι περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ ε, τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα προστατευμένα αυτά προϊόντα και περίπου 15 ε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια έχουμε από τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ποιότητα των γεωργικών μας προϊόντων είναι τμήμα των παραδόσεων, της διατροφής μας, του πολιτισμού μας, αλλά επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι η ποιότητα αυτών των προϊόντων μας δίνει ε, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και το προβάδισμα στις αγορές. Λοιπόν, θα πρέπει να επεκτείνουμε αυτό το κατάλογο προκειμένου να προστατεύσουμε και άλλα προϊόντα και να αξιοποιήσουμε την υψηλή ποιότητα των γεωργικών μας προϊόντων και στην παγκόσμια αγορά. Αυτό βέβαια περιλαμβάνει και την ανάγκη να προστατεύσουμε τα προϊόντα αυτά και στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με, με τις ΗΠΑ για το TTIP. Αλλιώς δεν θα είναι επωφελής ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντερσον. Αυτοί που στην Βρετανική κυβέρνηση εκπροσωπούν και τη Βόρεια Ιρλανδία και προωθούν το Brexit είναι ανεύθυνοι. Η Βόρεια Ιρλανδία γενικά ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι κοινοτικές ομάδες, ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, ε, διεθνή οικονομικά Ινστιτούτα ενισχύουν την περιοχή και βοηθούν έτσι ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις που θα δημιουργηθούν δυσάρεστες με τη συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας μετά την έξοδο. Οι γεωργοί μας επίσης ε, υπολογίζουν σε τεράστιες ε, ε, υποστηρίξεις και επιδοτήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να υπάρχει ένα σύστημα δίκαιο για την αμοιβή τους. Γι' αυτό λοιπόν η ευρωσκεπτικιστική δεξιά και η βρετανική κυβέρνηση θα αγνοήσουν την κατάσταση αυτή και το συμφέιν θα διαφωνήσει κάθετα. Ο κύριο Σεμπαστιά. Καλησπέρα σα. Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδε ε, άνθρωποι ε, διαδήλωσαν στη Βιγέρντε Κάνια, στην πόλη, στην Κουένκα, για να εμποδίσουν την ε, κατασκευή αποθήκη πυρηνικού υλικού. Σε ερώτηση που έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίστηκε ότι το σχέδιο αυτό δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες μελέτες ε, που υποχρεώνει συνθήκη Ευρατών, την οποία έχει υπογράψει και η Ισπανία. Και το Συμβούλιο Πυρηνικής Ασφάλειας καταγγέλει και πολιτικές πιέσεις και μάλιστα μελέτες με τις οποίες δεν συμφωνεί αυτό το Συμβούλιο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά και η θέση θεωρείται ε, ακατάλληλη από πολλούς εμπειρογνώμονες. Δεν θα πρέπει να μετατρέψει η, ε, Ισπανική κυβέρνηση τη Βιγέλντα Κάνιας σε πυρηνικό νεκροταφείο χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως τους πολίτες και χωρίς να έχει λάβει τα μέτρα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μια τόσο επικίνδυνη κατασκευή πυρηνικού υλικού και να μείνει αμέτωχη σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει αυτή η περιοχή χωματερή που δεν θέλει κανένας. Ο κύριος Μπάτεν. Ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε πως η Γερμανία δεν μπορούσε να αποστείλει Ούγκρους και λοιπούς Ευρωπαίους πολίτες ε, στις χώρες τους ε, εκτός εάν αποδείξει ότι οι φυλακές τους έχουν ανθρώπινες συνθήκες. Ε, προφανώς άμα δεν μπορούμε να αποστείλουμε αλλοδαπούς δεν μπορούμε να στείλουμε και Βρετανούς πολίτες σε ξένες φυλακές και έχουμε συχνά δει τις απάνθρωπες συνθήκες σε ελληνικές, ισπανικές και ουγγρικές φυλακές. Για να αναφέρω μόνο αυτά τα παραδείγματα. Θα απευθύνω τώρα επιστολή στην Υπουργό των Εσωτερικών για να αναστείλει τις εκδόσεις Βρετανών πολιτών σύμφωνα με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης σε ευρωπαϊκές χώρες όπου τίθεται ζήτημα συνθήκων στις φυλακές. Οπότε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή. Η Βρετανία χρειάζεται μια συνθήκη έκδοσης η οποία θα προστατεύει τους πολίτες μας σύμφωνα με το δικό μας δίκαιο και αυτό γίνεται μόνο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι τρελός ε, του Βοσπόρου, όπως ε, λέμε τον ε, Ερντογάν, ξαναχτύπησε. Τώρα ζήτησε από τον πρέσβη του να ασχοληθεί με ένα έργο της Συμφωνικής της Δρέσδης το οποίο ασχολείται με την ε, γενοκτονία των Αρμενίων για να μην ακουστεί η λέξη γενοκτονία. Ως μέλος της ε, Επιτροπής Πολιτισμού έχω να πω το εξής. Προτείνω στη Συμφωνική της Δρέσδης να διαγράψουν τη λέξη γενοκτονία και να την αντικαταστήσουν από την γερμανική συνώνυμη. Εμένα το Felkermord μου κάνει όπως και το Genocide ε, σημαίνει το ίδιο πράγμα. Όμως θα ήθελα να προειδοποιήσω την ε, τουρκική κυβέρνηση καθώς ε, κατεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά να κοιτάξει λίγο την ε, κατάσταση των Κούρδων η οποία αρχίζει και αυτή ξανά να μοιάζει με γενοκτονία και να σας πω επίσης πως δεν πρόκειται να ξαναπάω διακοπές στη χώρα αυτή. Κυρία Μέτσολε ta' faċli, ta' Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστα δίκτυα γρήγορου ίντερνετ. Πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης την καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χαμηλότερες τιμές. Δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα για τους παροχείς υπηρεσιών διότι είναι απαράδεκτο άλλα να διαφημίζουν σε σχέση με την ταχύτητα σύνδεσης και να μην ε, μπορεί ο πελάτης να χρησιμοποιήσει τις ταχύτητες αυτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή ενημέρωση για την ε, σωστή ταχύτητα, την πραγματική ταχύτητα, έτσι ώστε αυτά τα οποία συμφωνούνται να εφαρμόζονται. Το διαδίκτυο είναι κρίσιμο για τη ζωή μας σήμερα, εξαρτώμεθα από αυτό και γι' αυτό ζητώ να υπάρξει καλύτερη προστασία του καταναλωτή και χαμηλότερο κόστος. Από τον επόμενο χρόνο θα απαλλαγούμε από το roaming. Η πρόοδος αυτή θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και στον τομέα του διαδικτύου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε μια οικογένεια από τη Ρουμανία, του κυρίου Μπαντανάριου, που περνάει τα πάνδυνα από το προηγούμενο Νοέμβριο, κάτι που έχει προκαλέσει αγανάκτηση στη Ρουμανία και αλλού. Ε, φαίνονται να χρησιμοποιείται μέθοδη παρόμοια με αυτή τη ιερά εξέταση από την Ορβηγία και από την ε, υπηρεσία τη για την προστασία του παιδιού. Ε, η υπηρεσία αυτή κήρυξε του ε, γονείς ανίκανους να, να αναθρέψουν τα παιδιά τους με βάση τις θρησκευτικέ τους αξίες και τις πολιτιστικές τους αξίες ε, και ε, τους αφαίρεσαν ε, με τη βία τα παιδιά και τα ανέθεσαν σε μια ανάδοχο οικογένεια. Νομίζω ότι οι αρχές αυτής της Νορβηγίας παρερμηνεύουν την έννοια της προστασίας του παιδιού και παραβιάζουν τα δικαιώματα και των γονέων, την ιερή και απαράβατη ιδιωτική σφαίρα και το θεσμό της οικογένειας. Τα παιδιά είναι ένα θείο δώρο ε, και είναι απαράδεκτο ε, να εφαρμόζονται αυτές οι αντιχριστιανικές πρακτικές που καταστρέφουν τις οικογένειες στην Ορβηγία. Θα πρέπει να αναλυθούν δράσεις για να επανενωθεί επιτέλους η οικογένεια Μποντανάριου. Η κυρία Σμόκοβα. Σας ευχαριστώ. όπως όταν ταξιδεύουμε στις Βρυξέλλες ε, οι κύριοι Τούσκ, Γιούνκερ, Σούλτς χρησιμοποιούν ειδικέ πτήσεις. Δεν α, ε, ε, περνάνε αυτά που περνά ένας απλός πολίτης που προσπαθεί να ταξιδέψει και πρέπει να περάσει από 100 ελέγχους, από στρατιωτικούς, αστυνομικούς και αισθάνεται ανήμπορος και ανυπεράσπιστος και έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Αυτά θα πρέπει να σκεφτούν οι θύνοντες. Αυτό θέλουμε για τους συμπολίτες μας, ε, να περνάνε γολγοθα κάθε φορά που πρέπει να πάρουν αεροπλάνο. Ε, θα πρέπει κύριε Γιούνκερ, κύριε Σούλς, κύριε Τούς και εσείς που μπορείτε κάτι να κάνετε για να, βελτιώσετε, να βελτιωθεί η κατάσταση. Και οι πρόσφυγες από Συρία, Λιβύη και άλλες φτωχές αφρικανικές χώρες να μην έχουν λόγο να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους γιατί η παρουσία της αστυνομίας και του στρατού όχι μόνο δεν βελτιώνει την κατάσταση των προσφύγων, αλλά ίσα ίσα βοηθά στην έξαρση του εξτρεμισμού. Ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ. Ευχαριστώ. Ε, συνήθως ακούμε για τον Βλάντιμιρ Πούτινγκ στην αίθουσα όταν θέλουμε να επαναφέρουμε στην τάξη εκείνους ε, που κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για κάποια παλιδρόμηση που διαπιστώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάποια θεσμικά όργανα. Ε, και μάλιστα ε, όταν ε, η Ρωσία προσπαθεί να εξοντώσει τους Τατάρους και καταπατάει την ελευθερία της Κρυμαίας, τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας προσκάλεσε επίσημα τον Πούτιν για επίσκεψη στη χώρα του, στη Γαλλία. δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και να πιστεύω αυτά που είπαν για τα, για σήματα ε, μακραίων ε, παραδόσεων, αλλά για κάποια αρνητικά σήματα και μηνύματα που δίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για την ίση εργασία και το ίδιο και η κυρία Τάισεν. Οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό έχει γίνει αντικείμενο εγγύησης. Εμείς έχουμε όμως άλλο σύστημα διαφορετικού επίπεδου για καθηγητές, για νοσοκόμους κτλ. Και ιδιαίτερα οι νέοι καθηγητές, οι νέοι δάσκαλοι μου έστειλαν ένα mail και μου είπαν ότι αυτοί προσελήφθησαν μετά το 12 ε, κοστίζουν συνολικά πολύ λιγότερο από αυτούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι το 2011. Βέβαια δεν υπάρχει κοινοτικός νόμος ο οποίος να ε, περιγράφει τις κλίμακες των μισθών. Πάντως ε, δεν εφαρμόζεται η αρχή αυτή στην Ιρλανδία. Πώς μπορούμε να πούμε σε έναν τέτοιο καθηγητή που θα πληρώνεται τόσο λιγότερο ότι ο κοινοτικό νόμος προβλέπει τον σεβασμό της αρχής ίση αμοιβή, ίση εργασία. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε για την υπόθεση Μιλάμε για την υπόθεση ενός κοριτσιού που εξαφανίστηκε το 1977 και αυτός που θεωρείται υπεύθυνο για την εξαφάνιση του κοριτσιού αυτού παραμένει πάντα, ζει στην ίδια κοινότητα και δεν έχει δικαστεί ποτέ. Και κάποιοι τοπικοί πολιτικοί παρενέβησαν και αυτό οδήγησε σε μια απέσια κάλυψη της υπόθεσης από την Ιρλανδική αστυνομία. Εγώ έφερα τη δίδυμη αδελφή της Μέρη πέρυσι στο Κοινοβούλιο. Το άρθρο 2 δίδει το, καθιερώνει το δικαίωμα στη ζωή. Η Μέρη όμως των 6 ετών δεν μπόρεσε να χαρεί το δικαίωμα αυτό και δεν υπήρξε αναγνώριση του δικαιώματος της να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν υπήρξε έρευνα, επιτροπή έρευνας παρά παρά την, το αίτημα της νομικής ομάδας που ασχολήθηκε με την υπόθεση. Λοιπόν, η Μέρι Μπόιλντ έξι ετών προδόθηκε από το Ιρλανδικό κράτος. Ευχαριστώ κύριε Στερικάμπρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να, για να γίνει σεβαστό στο στόχο ε, του ελλείμματο. την περασμένη εβδομάδα η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από τις, από τις αυτόνομες κυβέρνησεις να αναλάβουν το σύνολο του, των εξόδων. Είναι ε, απαράδεκτο όμως και άδικο ε, να φυγοκεντρίζουμε το έλλειμμα. Γιατί ο καταλανικός προϋπολογισμός, για παράδειγμα, το 60% και παραπάνω αφορούν αυτό το κεφάλαιο. Και με τις περικοπές αυτές η Καταλωνία θα χάσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι σαν να κλείνει ένα χρόνο τα σοφρονιστικά ιδρύματα, τα δικαστήρια και τρία μεγάλα νοσοκομεία. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε ισορροπημένα τα δημόσια οικονομικά και του δημόσιου λογαριασμού, αλλά είναι απαράδεκτε οι περαιτέρω περικοπέ στην παιδεία ή στι κοινωνικέ υπηρεσίε. Γιατί λοιπόν η Ισπανική κυβέρνηση δεν μειώνει τι δικέ του δημόσιε δαπάνε στην άμυνα, για παράδειγμα, που είναι πάνω από 1% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Τι νόημα έχει ε, να κρατά Υπουργείο Πολιτισμού εφόσον οι ε, ε, αυτόνομε περιφέρειε είναι αρμόδιε για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Σήμερα ξενιστάμεθα και γανακτίζουμε για την ε, σύλληψη της Ολλανδέζας δημοσιογράφου ε, μετά από διαταγή του Ερδογάν. Ε, γιατί όμως η Ολλανδική κυβέρνηση δεν κάνει ε, τα ίδια και, και δεν κατηγορεί και τις ε, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όταν κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί ε, η Αμέρκερ δέχτηκε να διωχθεί δικαστικά ο κ. Μπάκερμαν. Επίσης, ε, πριν από μερικά χρόνια αναφέρθηκε, κατηγορήθηκε ο Λέχ Κατσίνσκι τότε ο πρόεδρος από, την, μια γερμανική εφημερίδα γιατί δεν τηρεόταν η ελευθερία του λόγου αλλά δυστυχώς υιοθετούνται δύο μέτρα και σταθμάκι. Γιατί δεν ε, υιοθέτησε ο κύριος ε, Σούλτς αρνητική στάση όταν έγινε η συμφωνία με την Τουρκία και τον κύριο Ερντογκάν. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστραφεί. Ο κύριος Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή πήγα στο Βελιγράδι για να παρατηρήσω τις βουλευτικές εκλογές. Είναι σημαντικό μήνυμα το ότι μια σαφής πλειοψηφία επέλεξε μια φιλοευρωπαϊκή πορεία για τη χώρα της. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα και οι επικοδομητικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες επέτρεψαν να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην περιφερειακή συνεργασία και στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία τώρα μπορεί να ασχοληθεί με την εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την εγγύηση της ελευθερίας των ΜΜΕ. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δύσκολους καιρούς και η φωνή της Σερβίας νομίζω θα μας βοηθήσει. Για να βοηθήσουμε τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία, εγώ θεωρώ πως ε, τα κεφάλαια 23 και 24 που αφορούν τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη θα πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκίλ. συγκλονίστηκα και εγώ όπως και τα 30 εκατομμύρια ΣΥΧ για την επίθεση στον ε, ναό που έγινε στην έση της Γερμανίας την προηγούμενη εβδομάδα και βεβαίως ε, θα ήθελα να απευθύνω τα συλληπιτήριά μου στους ε, τραυματίες. Καμία πίστη δεν πρέπει να στοχεύεται έτσι. Είναι ακατανόητο γιατί ριζοσπαστικοποιημένοι νέοι στοχεύουν αυτή την θρησκεία η οποία ταΐζει άστεγους και πεινασμένους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποθέτω ότι ο στόχος τους ήταν να σπείρουν την δυσπιστία. Πρέπει λοιπόν να βρουν, να ασχοληθούν τώρα με τους δράστες ε, οι γερμανικές αρχές ε, έτσι ώστε να καθισκάσουν τους ΣΥΧ ε, στο κρατήδιο της ΕΣΙΣ αλλά και οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη ότι η επίθεση αυτή θα αντιμετωπιστεί όπως και κάθε άλλη τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Πιμέντα Λόπεζ. Ευχαριστώ. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική παίρνουν πολύ δύσκολες και σημαντικές στιγμές. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας για να τεθεί τέλος σε, μια σε έναν επονίδιστο αποκλεισμό που ξεκίνησε από το 1976. Επίσης, ε, συνεχίζω, φτάσαμε σε, ένα, ε, σε μια κρίσιμη κατάσταση και στις συνευτικές διαπραγματεύσεις με την Κολομβία. Ε, κυρίως επειδή ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη έχει τις ΦΑΡΚ στον κατάλογο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. υποτίθεται ότι ε, γίνονται προσπάθειες δημοκρατίας, αλλά παρόλα αυτά κατηγορούμε την Βενεζουέλα και, άλλες και την Βραζιλία για τις προσπάθειες που κάνουν. Επίσης, στο σημερινό είχαμε ένα καταστροφικό ε, σεισμό με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες θύματα που χρήζει, χρήζουν άμεσης βοήθειας και υποστήριξης και οικονομικής και ανθρωπιστικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Ποσπίσιλ. Ευχαριστώ. Και εγώ κάτι παρόμοιο θέλω να πω με τον κύριο Στέφανετς. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχουμε με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επίτροπο, κυρία Γιώροβα, να θίξει αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Ε, μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια πολλών κρατών μελών για την κατάσταση. Στην Τσεχία μάλιστα η Τσεχική Βουλή αλλά και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας απέρριψαν την πρόταση της οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσο είναι απαραίτητες όλες οι οδηγίες, όλες οι διατάξεις της οδηγίας για να καταπολεμήσουμε την δρομοκρατία. μερικές ε, διατάξεις βρίσκονται εκεί απλώς για να ενοχλήσουν νόμιμους κατόχους ε, όπλων. Ο κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στις χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως στη Ρουμανία. Πρόκειται για την αρπαγή γεών από κερδοσκόπους που είναι μεταμφιεσμένοι σε αλλοδαπούς επενδυτές. Οι τιμές είναι εξευθυριστικές σε σχέση με άλλες χώρες, γι' αυτό και οι κερδοσκόποι ε, αρπάζουν, αγοράζουν σε εξευθυριστικές τιμές ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, εκτάρια, οδηγώντας σε ασφυξία τις μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε διακοπή των γεωργικών διαπραγματεύσεων. Έτσι, οι γεωργικές γεές αλλάζουν χέρια και χάνουν τη λειτουργικότητά της. Δεν καλλιεργούνται πια, παρά τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει την γεωργία και την, και την Δεν μπορεί να αγνοεί την κατάσταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι απαράδεκτη για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Δεχόφσκι. pane předsedající, jako vždycky jsem tady dneska zase poslední. Όπως τελευταίος μιλάω. Αλλά έχω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και το ξεχνάμε αυτό στη συζήτηση για την μετανάστευση, αλλά είναι σημαντικό. Είναι το θέμα της ψυχολογικής, της ψυχικής υγείας των προσφύγων. Άνθρωποι που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές που έχουν δει τους δικούς τους να πεθαίνουν αντιμετωπίζουν τώρα ακόμα χειρότερα πράγματα στην Ευρώπη. Γι' αυτό σας επαστήνω έκκληση κυρία Επίτροπε. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα και ένα από αυτά είναι το θέμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ωραία, ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Ε, η σύνοδο θα συνεχιστεί αύριο από τις 8.30 ε, το πρωί. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο την κυρία Βέροβα που ήταν παρούσα, μίλησε για όλα τα θέματα και ευχαριστώ.